και μεταρρυθμιστών έναν κατάλογο διορισμών που θα ενταχθούν στα, στα πρακτικά εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς τους διορισμούς αυτούς. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο 5η 9 του μηνός από τις 9 μέχρι τη 1, 3 με 5. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί και υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λύεται η συνεδρίαση.